Uh, Και τώρα περνάμε στην επόμενη συζήτηση στην ημερήσια διάταξη. Είναι η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου για το έτος 2013. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, κύριο Ντασίλβα Καλντέιρα. Θα ήθελα επευκαιρία να δώσω το λόγο λοιπόν πρώτα στον κύριο Δασίλβα Καλδέρα και ακολουθούν οι επόμενοι μιλητές. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο κύριε Σίλβα Καλδέρα. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσω αμέσως. Κυρίες και κύριοι, κύρια Αντιπρόεδρε Γεωργίευα, για μένα είναι τιμή η παρουσίαση της σας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δημοσιονομικό έτος 13 σε αυτή την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σημαντική στιγμή αλλαγής της Ευρώπης. Η Κομισιόν αντιμετωπίζει πολλές καινούργιες προκλήσεις και μία από αυτές είναι και η βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της άσκης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, στην αρχή αυτής της νέας αθαπανητικής περίοδου η ετήσια έκθεση του συνεδρίου λέει ότι δεν είναι ακόμη ικανοποιητική η δημοσιονομική διαχείριση της Ένωσης και οι διαχειριστές δεν είναι υπεύθυνοι μόνο για τη δαπάνηση των χρημάτων αλλά και για το ότι η δαπάνηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και είναι και αποτελεσματική. Όσον αφορά τη χρήση του προϋπολογισμού 148 δισεκατομμύρια πληρωμές έγιναν από τον προϋπολογισμό το 2013. Καταλήγουμε ότι αυτές οι δοσοληψίες το 2013 έγιναν όπως έπρεπε και επομένως έχουμε σχεδόν δώσει σε εισαγωγικά απαλλαγή. Αλλά παρά το ποσό, το ύψος αυτό των δαπανών υπήρξαν και άλλες υποχρεώσεις δημοσιονομικές για κατά 9 δισεκατομμύρια παραπάνω μέχρι και 322 μέχρι το τέλος του 2013. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση για τις χρηματικές ροές στην Ένωση και πρέπει να προετοιμάζεται τέτοια ροή για να προβλέπονται, να αποφεύγονται οι ελλείψεις χρημάτων και ρευστού. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι οι δαπάνες αυτές αφορούσαν πραγματικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη λιγότερο από το μισό των 14 δισεκατομμυρίων που πληρώθηκαν για εργαλεία δημοσιονομικού δημοσιονομικών διευθετήσεων δεν είχαν πληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ακόμη πληρωμές που δεν συμφωνούν με τους κανόνες. Θεωρούμε ότι το συνολικό λάθος, ποσοστιαίο λάθος για τις πληρωμές είναι 4,7% του 2013 μέχρι και 4,8% που ήταν το 12, με, από 4,8% που ήταν το 12. Και θεωρούμε ότι το 4,7% αυτό ετησίως είναι ακόμη υψηλό. Όλοι οι τομείς δαπάνων είχαν τέτοια υλικά λάθη, εκτός από τα 10,6 δισεκατομμύρια που δαπάνησε η Ένωση για την ίδια της τη διοίκηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το ποσοστό λάθους είναι μεγαλύτερο και το συμμερίζονται από κοινού οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να μειωθεί αυτό το ποσοστό λάθους και θα έπρεπε να είχε μειωθεί και να είχαν αποφευχθεί τα λάθη καταρχήν. Παραδείγματο χάρη το ποσοστό λάθους για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου μειώθηκε από 6,7% σε 2%. Θα μειωνόταν μάλλον εάν οι εθνικές αρχές είχαν χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που διέθεταν πριν υποβάλουν αιτήματα για πληρωμές στην Κομισιόν. Η πηγή του λάθους που θα έπρεπε να προσέξουν τα κράτη-μέλη είναι απαράδεκτα αιτήματα και σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων των δημοσίων προμηθειών. Κατ' εμάς, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, οι αρχές των κρατών μελών, πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στην αποφυγή καταρχήν του λάθους και μετά να τα διορθώνουν διότι έτσι τίθεται εν κινδύνο όλη η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής δαπάνησης. Κυρίες και κύριοι, η πραγματική περίοδος 7 με 13. Κατά την περίοδο αυτή βασίστηκε η Ένωση κυρίως στη δαπάνηση των διαθεσίμων χρημάτων και δεύτερον στην συμμόρφωση με τους κανόνες και μετά μόνο, και όχι πολύ, στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Έχουμε πολλά παραδείγματα στην έκθεσή μας από προηγούμενες εκθέσεις μας. 19 ειδικέ εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το 2013 για να δούμε πώς θα μπορούσαν αυτά να είχαν διορθωθεί. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν για αλλαγή από ήθη δαπάνη σε ήθη αποτελεσματικότητας. Αυτό θα σήμαινε κατά εμάς πρώτον μία πραγματική δέσμευση σε εθνικό και νοσιακό επίπεδο ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε. Δεύτερον, να τεθούν επαρκείς και σωστοί στόχοι για τα αποτελέσματα που ζητάμε και τρίτον και σημαντικότερον πρέπει να υπάρξουν τα σωστά κίνητρα για να επιβραβεύεται η αποτελεσματικότητα και να τιμωρείται η μη αποτελεσματικότητα. Μέχρι τώρα οι δημοσιονομικοί διοικητές της Ένωσης έπρεπε καταρχήν να δαπανίσουν τα χρήματα αλλιώς θα χανόταν. Και τέλος. Σημαντικό είναι επίσης τα αποτελέσματα από το ενωσιακό χρήμα να είναι και ορατά. Ιδιαίτερα θα έπρεπε η Κομισιόν να βελτιώσει την κάλυψη που κάνει της ετήσιας της αποτίμησης και της προόδου που θα έχει επιτευχθεί για την επίτευξη των στόχων του 2020. Πρόεδρε κυρίες και κύριοι, η βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης δεν είναι θέμα επιλογής μεταξύ δαπάνησης των χρημάτων, συμμόρφωσης με τους κανόνες και επίτευξης αποτελεσμάτων. Το θέμα είναι και τα τρία ταυτόχρονα. Έτσι ώστε ο προπολογισμό να γίνει πιο διαχειρίσιμος και με καθαρότερους κανόνες, στόχους και μεγαλύτερη απλότητα. Όπως δείχνει η έκθεσή μας, Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στην, να, να βοηθήσουμε το Κοινοβούλιο όσο και άλλα κοινοτικά όργανα για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντασίλβα Καλντέρα. Και τώρα εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπής το λόγο έχει η κυρία Γεωργίευα. Παρακαλώ. Thank you very much, Madam President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Καλτέρα, εισηγήτρια. Θα ήθελα να αρχίσω επαναλαμβάνοντας σε αυτό εδώ το χώρο το πόσο εκτιμούμε αυτήν την τόσο άρτια έκθεση που παρουσίασε το Ελληνικό Συνέδριο και πόσο επικοδομητικές είναι οι συστάσεις που διατύπωσε. Εντοπίσατε για το 2013 ε, ένα ποστό σφάλματος περίπου 7%. Ακόμα πάντως ε, απέχουμε αρκετά από το 2% του κατοφλίου το οποίο έχουμε θέσει ως ε, φιλοδοξία μας όμως βρισκόμαστε αρκετά πιο κάτω από εκεί που βρισκόμασταν πέρσι που είχαμε 4,8% και βεβαίως διαπιστώνουμε ότι η τάση η αυξητική των προηγουμένων ετών έχει αντιστραφεί. Γιατί φτάσαμε στο ρεκόρ του 148 δις ευρώ όσον αφορά την πρικοδότηση των προγραμμάτων που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπετε ευμένως ποια είναι τα αποτελέσματα των προσπαθειών που έχουν καταβάλει οι συνάδελφοι κατά τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τι συστάσει του ελεγκτικού συνεδρίου. Πάντω θα πρέπει να σα πω ποιο είναι για μένα το μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε. Είναι ότι θα πρέπει να επιμείνουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας. Κατά δεύτερο λόγο. Μα ενθαρρύνει πάρα πολύ το ότι, τώρα μπορούμε να βεβαιώσουμε όλο τον κόσμο ότι οι λογαριασμοί αυτοί τώρα δεν έχουν για 7η χρονιά τώρα επιτέλους ε, σφάλματα. Να, ποιο είναι το αποτέλεσμα, η καρπή του έργου που επιτελέσαμε και βλέπετε τι καταφέραμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε κάτω από το κατόφλι του 2%. Και θετική άποψη για όλε τι κατηγορίε δαπανών. Και είδατε μα τι γίνεται σε όλου του τομεί όπου έχουμε συνδιαχείριση στην, στην πολιτική συνοχή αλλά και στη γεωργία. Και επίση ετώνησα στην έκθεση, όπω και στο παρελθόν έκανα, για το ότι υπάρχει μια μεταβλητή που σίγουρα έχει επιπτώσει στην υπόθεση των λαθών. Ότι έχουμε πάρα πολύ περίπλοκους ε, ε, κανόνε όσον αφορά την επιλεξιμότητα, όσον αφορά τι δημόσιες προμήθειε, όσον αφορά τι δημόσιε ενισχύσει, Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπαθίε μας σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Εκεί όπου έχουμε πολλά προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε εάν θέλουμε να αποφύγουμε ε, την επιδείνωση κατάσταση στο μέλλον για να έχουμε καλύτερα σε επιδόσεις. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ε, κυρίους αξιωτικούς βουλευτές ότι ακόμα έχουμε κάποια προβλήματα που θα πρέπει να τα επιλύσουμε. Δηλαδή, τον πολίτη χαρακτήρα των προγραμμάτων μας και από την άλλη μεριά την ετήσιο χαρακτήρα των εκθέσεων του Ελληνικού Συνεδρίου γιατί πολύ συχνά γίνονται οι διορθώσεις αφορούν τις επόμενες χρήσει, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη τη χρήση και το έτος κατά την οποία δημοσιοποιείται η έκθεση. Να επομένω τι γίνεται με το ποσοστό σφάλματος, το ετήσιο και αυτό το οποίο λαμβάνεται υπόψη. Είδατε ότι είχαμε 2,2 ε, ρυθμό διορθώσεων, κάτι το οποίο μείωσε και θα μειώσει κι άλλο το ποσοστό σφάλματος. Δεν θέλω να πένευσε το σπίτι μου. Θέλω να κοιτάξουμε μπροστά. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε δύο πάρα πολύ ουσιαστικά σημεία. Πρώτα-πρώτα, ότι για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 έχουμε θεσπίσει νέε διατάξει και κανόνε ε, και λαμβάνει υπόψη τρει αρχέ, την ε, απλούστευση, την συρρήγνωση των διοικητικών δαπανών, ακριβώ όπω έχει πει το Ελληνικό Συνέδριο, να μην έχουμε πια τον κίνδυνο να πέσουμε σε περισσότερα ασφάλματα και επίσης να υπάρχει ευθύνη όσον αφορά τη συνδιαχείριση από πλευράς εθνικών αρχών, αλλά επίσης θέλουμε να υπάρξει και ανάλυση πολιτικής ευθύνης, πολιτικής ευθύνης σε εθνικό επίπεδο επίσης, κίνητρα να υπάρχουν κάποιες καθαρές ε, διορθώσεις μεσομικού χαρακτήρα, κάτι το οποίο είναι κίνητρο για ελέγχους και αυτό ακριβώ θέλουμε να γίνει για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Άλλο, δεύτερο σημείο ουσιαστικό είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πάρα πολύ σοβαρά την σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις επιδόσεις μας και αυτό να είναι το κυρίαρχο πνεύμα και αυτό θα αποτελέσει για μένα το σημείο που θα εστιάσω την δράση και την πολιτική μου. Τα έχουμε πει αυτά με τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έχουν υπόψη τα κράτη-μέλη και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι. Πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε πάρει πάρα πολύ σοβαρά την σύσταση που διατυπώσατε ότι θα πρέπει να συγκροτήσουμε ένα διοργανικό γκρουπ, μια διοργανική ομάδα εργασίας οπότε αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οι Ευρωπαίοι έχουν προσδοκίες από μας. Θα πρέπει να τους αποδείξουμε ότι προστατεύουμε τα χρήματα τα οποία εισφέρουν και ότι τα χρησιμοποιούμε για το συμφέρον εκείνων. Πρόεδρε Καλτέρα. θεσμευόμαστε πάρα πολύ σοβαρά να συνεργαστούμε με το Ελληνικό Συνέδριο κατά διπλό τρόπο με την συμμόρφωση και με τις σωστές επιδόσεις που οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα ε, αρχίζει η συζήτηση με πρώτη την εισηγήτρια, κυρία Γκρέσλε. Ε, ε, πρόεδρε, κύριε Καλδέρα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Το πιο ανησυχητικό σε αυτή τη μεγάλη έκθεση είναι τα αποτελέσματα είναι σε τρίτη θέση. Το σημαντικότερο είναι οι δαπάνες. Μα κυρία Επίτροπε, αν καταφέρετε αυτό να το καταπολεμήσετε θα είστε ηρωίδα μου. Γιατί εγώ φοβούμαι ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως είχε. Το έχω ακούσει δέκα φορές ότι όλα θα λυθούν και θα αλλάξουν με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, με τις νέες ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Ανεργία των νέων, τι κάναμε για την καταπολέμηση. Ε, ένταξη των Ρωμά, τι καταφέραμε. Αντί να τα πούμε αυτά, ε, τσακωνόμαστε γιατί δεν έχουμε αποτελέσματα και ε, ταλανιζόμαστε και αναλωνόμαστε με ε, τα σφάλματα. Έχω πολλές ερωτήσεις. Γιατί στα περιφερειακά ταμεία έχει τόσο μεγάλες διαφορές το ελεγκτικό συνέδριο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2,8 και 6,9 ή στην ανάπτυξη της υπαίθρου 5 και 19 λέει η Γεωργία και το ελεγκτικό συνέδριο 6,7. Γιατί γίνεται αυτό. Είναι σύγκρουση συμφερόντων, θέλουν κάποιοι να προστατευτούν από δικαστικές εισαγωγές. Έχω πολλές ερωτήσεις, χρηματοδοτικά μέσα. Γιατί μόνο 47% φτάνουν στους τελικούς δικαιούχους και ε, καταπολέμηση της απάτης. Είναι λυπηρό όταν ε, έχουμε μια υπηρεσία που δεν είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Επίσης υπάρχουν και λανθασμένα στοιχεία που δίνουν οι κρατικές αρχές. Στις αιτήσει εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών ε, βλέπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πολλές διορθώσεις. Όπως και στην Ευρωζώνη, μήπως χρειαζόμαστε και εδώ ε, κυρώσεις για λανθασμένα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία ε, Κρέσλε, η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίσατε κυρία Γεωργίευα ε, στο νέο χαρτοφυλάκιό σας και ευχαριστώ πολύ κύριε Καλδειρα ε, για τις προσπάθειες που κάνετε για τα νέα σχέδια, τις νέες αναλύσεις και τις νέες προτάσεις που είναι και σοφές και αξιόλογες. Έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα νέο κοινοβούλιο και μια νέα δημοσιονομική περίοδο και με την ίδια κρίση που διονύζεται εδώ και 7 χρόνια και είναι βιβλική καταστροφή ναι. από τις πληγές, τις βιβλικές. Ε, όλο και περισσότερα έχουμε προβλήματα ε, με πληρωμές. Αυτά είναι πρωτοφανή προβλήματα. 300 δις τώρα μας τάζει ο κύριος Γιούνκερ για επενδύσεις, αλλά με κάποιες κατασκευές περίεργες οικονομικές ε, και το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο μας λέει προσοχή και κυρία Γεωργέβα χρειάζονται αυτά εποπτεία. Και ο έλεγχος ε, των ε, μέτρων που έχουμε, που είναι όλο και πιο δύσκολα κάθε φορά και χρειάζεται συνεργασία με τις οικονομικές αρχές. Και νέα καμπανάκια που χτυπάνε για τους ιδίους πόρους, το ελεγκτικό συνέδριο μας λέει ότι υπάρχουν προβλήματα αξιοπιστίας για το πώς υπολογίζεται το ΑΕΠ του κάθε κράτους και κάθε φορά έχουμε μεγαλύτερα ελλείμματα και χειρότερο έλεγχο στα σύνορα, οπότε χάνουμε και από και ιδίω πόρους. Ανησυχούμε πάρα πολύ, όχι μόνο για τις δαπάνε, αλλά κυρίως και για τα έσοδα. Εν ευχαριστώ τον κύριο Καλδέιρα και το ηλεκτρικό συνέδριο που εντόπισε αυτά και τι εξοδέψαμε στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για το 290 ε, ευρώ ανακάτοικο και αναέτος. 290 ευρώ είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Και ο πραγματικός ουσιαστικός ε, βαθμός φαλμάτων είναι μόνο 13,6 ευρώ ανακάτοικο και έτος. Μπορεί να φαίνεται λίγο αυτό, αλλά είναι αρκετό για να χρειαστεί μελέτη και μεγαλύτερο έλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, ε, σας ευχαριστώ και πάλι που το ελεγκτικό συνέδριο κάνει αυτή τη ε, δουλειά και μετά και τις τάσεις και τα μεγέθη. Καλά, τα 45 δις της Γεωργίας ε, μειώνεται εκεί το σφάλμα κατά 0,2 ενώ στην ανάπτυξη της υπαίθρου αυξάνεται. Είναι λιγότερα τα χρήματα αλλά το σφάλμα είναι σχεδόν διπλάσιο, 6,7. Δηλαδή κοιτάμε και τα μεγέθη και τις τάσεις, αν αυξητικές ή αν μένουν μειούμενες. Ε, θα ακολουθήσουμε τη σύσταση ε, του ελεκτικού συνεδρίου να είμαστε στραμμένοι προς μια κουλτούρα αποτελεσμάτων, αλλά με κίνητρα. Όχι κάθε φορά να ψηρίζουμε τις δαπάνες που μειώνονται ε, και αυτό αυξάνει και τα προβλήματα και τη δυσφορία των πολιτών και των διοικήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσαρνέσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καρδίρα και τον κύριο Λάζαρο από το ελεγκτικό συνέδριο. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί δεν είμαστε εδώ σε ακρόαση αλλά στην Ολομέλεια με παρουσία της κυρίας Γεωργίευα στο Newsweek αυτής της εβδομάδας δημοσιεύεται ένας χάρτης που δείχνει τα προβλήματα των διαφόρων υπήρων και για την Ευρώπη το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανεργία των νέων. Και δαπανούνται χρήματα για προγράμματα καταπολέμησής της, αλλά όχι και πολύ σωστά μου φαίνεται όχι πολύ αποτελεσματικά τουλάχιστον. Είναι καλό που η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου θέτει το πρόβλημα της αποτελεσματικότητας. Η διαχείριση των πόρων της Ένωσης δεν γίνεται σωστά. Πρέπει να βελτιωθεί. Να βελτιωθεί. 322 δισεκατομμύρια και αναμένεται ότι η Ευρώπη θα δημιουργεί όλο και περισσότερα χρέη. Ο, τα ποσοστιαία λάθη που σημειώθηκαν είναι λίγο χαμηλότερα από παλαιότερα, παραμένουν και πέρσι και φέτος λίγο κάτω από το 5% και οι πιο προβληματικές περιοχές είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου και η πολιτική της συνοχής είναι δηλαδή οι τομείς όπου, όπου λέγω, οι νέες και πτωχότερες χώρες της Ευρώπης είναι πιο ευάλωτες. Ευχαριστώ. κύριος Αλή έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμε Αντιπρόεδρε της ε, Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε Καλτέρα, θα ήθελα να συγχαρώ το ε, ελεκτικό ε, συνέδριο για την ετήσια αυτή τελετή κατάθεσης και παρουσίασης της έκθεσης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα σωστό που να εκτιμά και να υπολογίζει το ΑΕΠ των κρατών μελών για να υπολογίζονται και ήδη οι πόροι που είναι το 70% του κοινοτικού προϋπολογισμού. Τονίζω τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στις επαληθεύσεις ε, και στις αναφορές και στην υποβολή των εκθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της δεν συμφωνεί με τους υπολογισμούς πολλές φορές του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά μου φαίνεται ότι έχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις σχεδόν για τα πάντα. Ε, μακροοικονομικά και λογιστικά και έχω και αμφιβολίες. Είδα την ε, αρνητική εκτίμηση ε, του ΑΕΠ, της αντίστοιχης ομάδας δηλαδή και ε, είδα και τις στατιστικές που δίνονται από τους θεσμούς υπάρχουν διεθνή Ινστιτούτα που βγάζουν μελέτες το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θεσμία, ε, οργανώσεις, η Παγκόσμια Τράπεζα, δεν μπορούμε να δανειστούμε και από αυτές τις πηγές κάποια στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, τα αρνητικά υπάρχει και κάτι θετικό. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σημασία των συστάσεων και συμφωνεί να τι εκτελέσει. Η εκτέλεση του προπολογισμού και ο λογιστικό έλεγχο θα πρέπει να βασίζονται σε αποτελέσματα και αν ε, έχουν επιτευχθεί οι βασικοί στόχοι και μόνο έτσι βελτιώνεται ο προπολογισμό. Με συντονισμό των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα τη διοίκηση του κράτου, τοπικό, περιφερειακό, κρατικό από την αρχή των προγραμμάτων. Θα πρέπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βοηθήσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Στάς. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, κυρία Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα γεγονότα είναι οδυνηρά για μας, το είπανε και οι συνάδελφοι. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι το 80% είναι στην συνδιαχείριση, στην υπευθυνότητα με τα κράτη-μέλη. Εκεί είναι τα προβλήματα. Τα κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Το είπε ο κύριος Καλντέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ξέρουν τα κράτη ότι γίνονται σφάλματα, δεν κάνουν τίποτα. Το ποσοστό των σφαλμάτων στην ανάπτυξη πέθρου, την αλληλεία, ε, στην υγεία 6,7% και στο περιβάλλον. Πρέπει να φτάσουν στο 2%. Εγώ προσθέτω ενέργεια, μεταφορές, περιφερειακή πολιτική. Τώρα 9% επεμβαίνουν τα κράτη-μέλη και γίνεται αυτό ως διαμαγείας 3,9. Απασχόληση και κοινωνικά 3,1 μπαίνουν τα κράτη-μέλη και βγαίνει 1,8. Επεμβαίνουν τα κράτη-μέλη αλλά χρειάζεται πρόγραμμα δράσης υπό την ηγεσία της κυρίας Γεωργίευα και τελικά να υπάρξει και μια εθνική δήλωση ε, των Υπουργών ε, δήλωση αξιοπιστίας και στα ομοσπονδιακά κράτη αυτό είναι συνδυασμός και των ομοσπονδων κρατηρίων και των αντιστοίχων υπουργών οικονομικών. Και ε, υπογράφει ο υπουργό, λέει έχω κάνει τη δουλειά μου, έχω κάνει τον έλεγχο, υπάρχουν κάποια σφάλματα και αν δεν γίνει αυτό τότε θα πρέπει να φέρει την ευθύνη ο εκάστοτε υπουργό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάλλη. Sì, grazie Presidente. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κάτι να σας πω όσον αφορά αυτές τις ε, υποδείξεις του Ελληνικού Συνεδρίου. Για αυτή τη θητεία θα πρέπει να μου πείτε ποια είναι η προσθεμένη αξία που πρόκειται από τα προηγούμενα χρόνια. Ε, έχουμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις, έχουμε ε, τα διάφορα προγράμματα και οπότε η έκθεση αυτή μας δείχνει το πώς τα κρατημέλη μπορούν να εγγυηθούν και αποτελέσματα για τη χρηματοδότηση. Γιατί ακριβώς αυτό το οποίο θέλουν τα κρατημέλη είναι το να διασπαρίζουν αυτά τα χρήματα. Δεν σέβονται τους κανόνες και τελικά αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει είναι να έχουμε κάποια αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων. Οπότε η διασπάθηση τόσων εκατομμυρίων που προέρχονται από αυτού που κάνουν κάποιε θυσίε και πληρώνουν του ε, φόρου του και από την άλλη μεριά να έχουμε τέτοιε φορολογικέ ε, αδικίες. Όλα αυτά είναι αχρίαστα, όλα αυτά είναι επιζήμια Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει διαχείριση από πολλά μελών των σχετικών κονδύλων. Οπότε για πετε μας, πώς γίνεται, αν μπορούμε να δούμε τι γίνεται, αντί να έχουμε μια πολιτική που να βοηθάει τον Ευρωπαίο, τελικά αυτό το οποίο κατησχεί είναι τα ε, συμφέροντα εκείνων που έχουν το χρήμα. Αυτό δεν είναι σωστή διαχείριση. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Βαϊλή. Βιλίμσκι, ευχαριστώ. Εγώ διερωτώ με Πώς μπορούν ανερυθρίαστα ορισμένοι να μιλούν εδώ μέσα. Ο κύριος Γιούνκερ έκανε φορολογικό παράδεισο τη χώρα του και από την άλλη οι πληθυσμοί της Ευρώπης ε, δυνοπαθούν και έρχονται να συγχρηματοδοτήσουν αυτά που έκανε στη χώρα του ο κύριος Γιούνκερ. Και από την άλλη ερχόμαστε και συζητούμε για 7 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακάλυψε ευτυχώ το ελεκτικό συνέδριο, που το 4% των πόρων είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και παρατύπως. Και ποιος αναλαμβάνει παρακαλώ ποια ευθύνη αυτοί που είναι απόντες και είναι τώρα στον πάρτο βουλευτών θα αναλάβουν την ευθύνη για τα 7 Ποιος είναι υπόλογο σε πάση περιπτώσει. 120 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν το 1 τέταρτο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλούνται από τη φτώχεια. Και δεν υπάρχει δυνατότητα με πόρους τη Ευρωπαϊκής Ένωσης των φορολογουμένων να γίνεται αυτή η διαχείριση συμπέρασμα να ξαναγυρίσει σε κρατικό επίπεδο η ενίσχυση γιατί μόνο οι ίδιες οι χώρες ξέρουν τι γίνεται στην επικράτεια, πώς πρέπει να δαπανηθούν τα λεφτά και πώς θα ελέγχονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα προσπαθήσουμε να σεβαστούμε όλοι το χρόνο ομιλίας μας, ο κύριος Σαβαρμά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και το συγχαίρω η ετήσια έκθεσή του για το 2013 ρίχνει περισσότερο φως στην κατάσταση. Το ποσοστό λάθος ήταν 4,7% και λέει ότι ε, θα μπορούσε να ήταν 6,3 αν δεν είχαν ληφθεί ορισμένα μέτρα, τελείως απαράδεκτο. Αλλά το θέμα είναι η ποιότητα, όχι η αριθμή. Ένα παράδειγμα της αξιοπιστίας αυτών των πληροφοριών που δίνουν τα κράτη-μέλη στην Κομισιόν. Στη διαθροτική πολιτική το ποσοστό λάθους σύμφωνα με την ε, Κομισιόν είναι μόνο 2,8%. Περιμένετε όμως. Άμα δούμε τα πράγματα πιο καλά βλέπουμε ότι είναι 6,9% κατά το ελεγκτικό συνέδριο. Μια από τις πιο σημαντικές παρατηρήσεις του λοιπόν είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εθνικές αρχές στα κράτη-μέλη είχαν επαρκείς πληροφορίες. Κύριε Πρόεδρε, αυτά πρέπει να διορθωθούν. Ο δημοσιονομικός έλεγχος πρέπει να γίνεται από πάνω μέχρι κάτω σε όλα τα προγράμματα και για να γίνει αυτό χρειάζεται πλήρης διαφάνεια και πλήρης χρήση όλων των πληροφοριών που διαθέτουμε. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτά που είπε η Επίτροπος Γεωργίευα Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε ο χρόνος σας. Τελείωσε ο χρόνος σας. Όχι, τελείωσε ο χρόνος σας. Με συγχωρείτε. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπόχουσλαβ Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Καλτέρα. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ. Για πρώτη φορά τώρα βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα που εγκλίνεται από ένα νέο κοινοβούλιο και από τόσους νέους συναδέλφους. Οπότε θα πρέπει να ε, πω ότι έχουμε και καινούργια επιτροπή, οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το μήνυμα, θα πρέπει να κλείσουμε έτσι αυτόν τον κύκλο ε, τον εκπαιδευτικό, γιατί είπαμε ότι κάποια μέλη κάνουν συνεχείς βελτιώσεις και είναι κάτι αυτό το οποίο χρειάζεται διότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να δουλεύουμε με σοβαρότητα και με συνέπεια και όχι να επιδιώκουμε τα πρωτοσέλιδα και τους πηχαίους τίτλους. Επομένως, δεν ε, πρόκειται εδώ περί κάποιου αυτού σκοπού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το έργο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Θα πρέπει κατά αυτή θητεία να δουλέψετε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αλλά επίσης θα πρέπει να έχετε ξεκάθαρο στόχο μπροστά σας. Και έτσι θα πρέπει να πετύχετε τους στόχους αυτούς που έχουμε θέσει είναι τόσο σημαντικοί. Κυρία Επίτροπε Γεωργίευα και εσείς αλλά και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας θα πρέπει να έχετε τα μέσα στη διάθεσή σας για να μπορέσετε να αποτιμήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο και τις υπόλοιπες συνέπειες των κοινωνικών προγραμμάτων και τα κρατημέλη και οι περιφερειακές αρχές επίσης ε, ε, είναι συνεργάτες σε αυτό και θα πρέπει όλοι να διασφαλίσουμε ότι κάθε δεκάρα της κοινοτικής χρηματοδότησης αξιοποιείται, πιάνει τόπο και να μην ξεχνάτε ότι πρέπει κανείς να επενδύει, όχι να ξοδεύει. Να συζητήσουμε πώς μπορούμε στους διάφορους τομείς να έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Θα πρέπει να συγκροτηθεί αυτή η διοργανική ε, ομάδα εργασίας για τις επιδόσεις μας και θα πρέπει να παρακολουθούμε εδώ πλευράς Κοινοβουλίου όλους τους τομείς πολιτικής και έτσι να μπορέσουμε να ε, έχουμε λήψη για το τι είναι επιδόσεις στην χρηματοδότηση των ε, ε, προγραμμάτων. Βίστησεν, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι το Ελληνικό συνέδριο πολλές φορές δεν εγκρίνει κάποιου λογαριασμού γιατί υπάρχουν τόσα λάθη που είναι πολύ παραπάνω από το κατόφλι του 2%. Αυτό το ξέρετε, δεν σας λέω τίποτα καινούργιο. Οπότε να σας πω κάτι άλλο. Να σας πω ότι από τη μία μεριά δεν έχουμε ενωσιακή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις δαπάνες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το ότι έχουμε τόσο μεγάλο προϋπολογισμό αλλά δεν θεωρούμε ότι τα χρήματα πιάνουν τόπο. Θα πρέπει τα χρήματα να πάνε στα κράτη-μέλη και εκεί να αξιοποιούνται. οι υποσχέσεις υπερκαλύπτουν τα όσα διαθέτουμε. Πρόκειται για μια βόμβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει αυτό να το δούμε στα σοβαρά. Αλλιώ θα αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικά προβλήματα στο μέλλον. Παρακαλώ αυτό λάβετε το υπόψη σοβαρά. Αυτό είναι το μήνυμά μου το σημερινό. Άρνοτ, ένα λεπτό. Δεν, δεν αρκεί 60 δευτερόλεπτα για να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση που δείχνει την κακοδιαχείριση. Εδώ βλέπουμε σκάνδαλα να περιγράφονται με πολυεθνικές, με ψεύτικες, ε, με αγροτικές επιχειρήσεις κτλ. Πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Κάθε φορά που ε, φτωχεύει ένα κράτος μέλος, φτωχεύει όλο το σύστημα. Υπάρχουν ακόμα 3,7% ποσοστά λάθους. Πέρυσι η Κομισιόν απλώς αγνόησε ότι το 21% των συστάσεων των ελεγκτών το σε, είχαν εφαρμοστεί λίγο ή πολύ. Αν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έκαναν κάτι τέτοιο θα φυλακίζονταν και αν υποβάλλονταν λανθασμένοι λογαριασμοί. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Αλιό για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο για τη σαφήνεια της έκθεσης αυτής. Η χρηματική και η οικονομική διαχείριση στην Ένωση δεν ήταν πάντα ικανοποιητική. Η Ένωση δαπανά τον προϋπολογισμό με βασική ανησυχία να δαπανίσει για τη δαπάνη, χωρίς να την νοιάζει αν πιάνουν τόπο και πού πάνε τα λεφτά και τι συνέπειες έχουν αυτά. Ε, επίσης σημειώνουμε τις δαπάνες που ε, γίνονται παράτυπα ε, ε, ε, με κάποια σεμνότητα τα ονομάζει σφάλματα, αλλά είναι απάτη. Ε, το πρόβλημα της διαφθοράς είναι αυτό σε κάποια έργα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ερχόμαστε να προσθέσουμε και τις ε, υποχρεώσεις ανεξόφλητες που είναι 322 δις ευρώ περίπου και θα καταλάβετε γιατί όλο και λιγότεροι πολίτες πιστεύουν σε αυτό το σύστημα. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο συγκλονιστική γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπαγορεύει τι θα κάνουν κυρίαρχα κράτη ενώ δεν μπορεί η ίδια να βάλει τάξη στον οίκο της. Για 1,5 λεπτό το λόγο ο κύριος Ντόιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου, κυρία Γεωργίευα, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς το Ελεγκτικό Συνέδριο για την έκθεση που έχουμε ενώπιον μας. Δεν συμφωνώ με τους συναδέλφους μου που διαφώνησαν με την έκθεση. Είναι μια καλή η έκθεση που βοηθάει το Κοινοβούλιο να βελτιώσει τις εργασίες του. Θέλω να σας θυμίσω τα δύο βασικότερα στοιχεία που επανέλαβε εδώ για μας ο κύριος Καλτέρα. Το 2014 ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 148 δις δαπάνες εκ των οποίων 4,7% δεν ήταν σύμφωνα και συμμορφούμενα με τους κανόνες. Και η κατηγορία σφάλματα λοιπόν κάλυπτε περίπου 7 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία και ε, αυτό σημαίνει για μας πολλή δουλειά για να τα διορθώσουμε τα σφάλματα και τα προβλήματα. Υπάρχει όμως ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν συζητούμε πολύ συχνά εμείς εδώ. Και αυτό είναι το ε, Τα 7 δι ε, αυτά των σφαλμάτων μπορούν να συγκριθούν με τα 25 ε, και μισό δισεκατομμύρια που δεν καταβάλλονται για την πολιτική συνοχή. Δηλαδή, ο κοινοτικός προπολογισμός δεν είναι σωστός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόν. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και το ελεκτικό συνέδριο και νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ δέχονται ότι ακόμα μια φορά μας είπε το συνέδριο ότι ήταν τακτικοί οι λογαριασμοί αν και πολλά ακόμη πρέπει να διορθωθούν για τις πληρωμές. Το ποσοστό λάθος 4,7% είναι πολύ ψηλό. Και θα ήθελα να πω όπως και οι άλλοι ότι εδώ μιλάμε όμως για λάθη, όχι για απάτες. Επίσης, τα περισσότερα από τα λάθη γίνονται σε επίπεδο κρατικό και υπάρχουν αριθμοί που δείχνουν ότι το ποσοστό λάθους είναι πολύ ψηλότερο από, στα κράτη-μέλη από ό,τι στα προγράμματα που τα διαχειρίζεται η απευθείας η Ένωση. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη, ιδίως αυτά που αποδεικνύονται προβληματικά κάθε χρόνο, να κάνουν κάτι Πώς θα μπορούσαν λοιπόν τα κράτη-μέλη να μειώσουν το ποσοστό λάθους τους. Όπως και άλλοι λοιπόν θα ήθελα να τονίσω το θέμα της αποτελεσματικότητας. Αγαπητέ συνάδελφε, τελείωσε ο χρόνος σας. Σας παρακαλώ να τελειώνετε, να σε καταλήγετε. Έλεγα ότι είχατε τελειώσει το χρόνο σας, αυτό σας έλεγα. Καλά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο κύριος Άσχορθ για ένα λεπτό. Πρόεδρε. Ενθαρρύνθηκα πάρα πολύ από τη θετική στάση των ελεγκτών και της Επιτρόπου. Πολύ σωστά είπαν και οι δύο ότι πρόκειται για μια νέα αρχή, για ένα νέο ξεκίνημα και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να λύσουν επιτέλους χρονίζοντα προβλήματα. Ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στο θέμα μιας αλλαγής ηθών, συμφωνώ. Αλλά προτείνω να αρχίσουμε αυτή την αλλαγή ηθών από εδώ, από το Κοινοβούλιο. Γιατί εμείς είμαστε οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των λαών. Εμείς είμαστε το Κοινοβούλιο που ζήτησε πρώτη φορά διαφάνεια για τους πολίτες. Αλλά δεν έχουμε δικαιοδοσίες για να καθορίσουμε τον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε δικαιοδοσίες για να ελέγξουμε τις δαπάνες και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για να μπορούμε να μετράμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι δαπάνες. Μόνο τότε αν έχουμε τέτοιες δικαιοδοσίες θα μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε τα ήθη. Ευχαριστώ. Κυρία Αντινόλφη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Συνεδρίου για την έκθεσή σα. Μένα με σοκάρει αυτό το ποσό σφάλματο που συνεχώ αυξήθηκε το 2009. Νομίζω το πρόβλημα ε, αφορά 30 Ε, Είναι κάτι δομικού πια χαρακτήρα, διωτικού χαρακτήρα. Είναι κάτι το οποίο αφορά την ευρωπαϊκή διοίκηση. Έχουμε α πούμε τις ε, συντάξεις, κάποιε αποζημιώσει ε, άλλες ε, δαπάνες φορούν τα ακίνητα. Τι γίνεται. Σε μια τέτοια συγκυρία ιστορική που έχουμε την κρίση που ζητάμε τόσο από τους Ευρωπαίους θα πρέπει να ασκούμε έναν έλεγχο πάρα πολύ προσεκτικό για οποιαδήποτε δημόσια σύμβαση, προμήθεια, δαπάνη. Ε, το ίδιο ισχύει και για όλα τα οικοδομήματα, όλα τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ θα πρέπει να προσέξει και να βελτιώσει όσο είναι δυνατόν ε, τα όσα γίνονται στο Λουξεμβούργο πλευρά τη φορολογική. Ο κύριος Μπονάνο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αρχίζω με ευχαριστίες και να χαιρετήσω και τους δημάρχους που έχουν έρθει εδώ από το Πεδεμόντιο, Ιταλοί δήμαρχοι ε, στο θεωρείο των επισήμων με συνοδεύουν και ε, είναι οι δήμοι και οι κοινότητες η ε, αφετηρία της δημοκρατίας και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή και στην πρωτοπορία. Είναι η αφρόκρεμα των Ιταλικών θεσμών. Έχω ένα λεπτό, τι να πεις ένα λεπτό. Στην εμπειρία μου ε, ως βουλευτής ε, βοήθησα στην καταπολέμηση της μαφίας και ε, συνήθισα και τον Πέτρο Γκράσο που ήταν εισαγγελέας κατά της μαφίας και τώρα είναι πρόεδρος της Γερουσίας και μου είπε ότι έχει αλλάξει η μαφία δεν ήταν ο νονός όπως ήταν η ταινία, η Σικελία και τα λοιπά τα κλισέ που ξέρετε στην Νότια Ιταλία τώρα η μαφία πάει εκεί που είναι τα λεφτά και που είναι τα μεγάλα συμφέροντα Γι' αυτό ακούω για τα 7 δισεκατομμύρια του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι εδώ η μαφία και στο Λουξεμβούργο. Παντού έχει πλοκάμια. Συμμετέχει σε όλες αυτές τις δραστηριότητες ε, που ε, ε, όλα αυτά τα απεχθή πράγματα που βλέπουμε και είναι ταυτόσιμα με την Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Σμιτ για 1,5 λεπτό. Η έκθεση ε, για το 2013 μας λέει 4,7 ποσοστό σφάλματος. Χωρίς τις ε, διορθώσεις ε, θα έφταναν και το 6,3%. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος μειώθηκε κατά 0,1%. Παρ' όλα αυτά 6,3% είναι χρήματα που έχουν δοθεί σε λάθος δικαιούχους το ελεκτικό συνέδριο ε, είπε ότι θα πρέπει να ελέγχονται ως προς τις παρατυπίες πάντα οι εκτελέσεις των προπολογισμών και ε, είναι ανησυχητική εκ των προτέρων έλεγχη. Κανονικά θα πρέπει να εντοπίζονται ε, νωρίς αυτά τα πράγματα, να αποκαλύπτονται και να διορθώνονται πριν καταβληθούν τα χρήματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η κατάσταση είναι αφόρητη. Θα πρέπει να δοθούν μηνύματα ε, και οι μηχανισμοί ελεκτικοί που διαθέτουμε να ενισχυθούν και να εφαρμόζονται σωστά. Είναι η 20η αυτή η εκτήσια έκθεση και πραγματικά τρομακτική η εκθεση και κρίμα τα κράτη-μέλη μετά από 20 χρόνια ελέγχων, διορθώσεων, υποστήριξης του ελεγκτικού συνεδρίου ακόμα δεν έχουν καταφέρει να κάνουν χρηστή διαχείριση και δεν μπορούν χωρίς σημαντικό σφάλμα να δαπανούν τα χρήματα. Είναι χρήματα των φορολογημένων. Αυτό μας βλάπτει. Όπως ο καθένας φροντίζει τα ιδιωτικά του οικονομικά και έχει χρηστή διαχείριση, θα πρέπει το αντίστοιχο να συμβαίνει σαν καλός οικογενειάρχης και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνο με τις γενικές ευχαριστίες προς το ελεκτικό συνέδριο, είδαμε ότι το ποσοστό σφαλμάτων στην εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού το 2013 έχει πέσει λίγο σε σχέση με το 4,8 πρόπερση. Μα μόνο αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο αναφορά τι έγινε το προηγούμενο έτος. Όχι, όποιοι ξέρουν τι γίνεται με τα κοινοτικά κονδύλια ξέρουν ότι διαφέρει καμπύλη των δαπανών. Στην αρχή είναι λιγότερες οι πληρωμές και όσο ολοκληρώνονται και εγκρίνονται έργα των κρατών, τόσο μπαίνει το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν που ήμασταν πριν από 7 έτη, ε, στο ίδιο χρονικό σημείο ε, της περίοδου 2000-2006. Και τότε ήταν 7,3% το ποσοστό σφάλματος. Με άλλα λόγια, ε, σήμερα μετά την προγραμματική περίοδο 7-13 έχει μειωθεί κατά 2,6 ε, ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη επταετία. Και είναι νομίζω αυτό πολιτική επιτυχία. Από εκεί και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα σφάλματα. Ε, το κλειδί είναι τώρα στα κράτη-μέλη και παραθέτω από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί χρειάζεται αυτό για μερικούς συναδέλφους, καμιά φορά παραθέτουμε ε, το πρωτότυπο κείμενο. Παρά τις υψηλές παρατυπίες και σφάλματα, οι κρατικές αρχές έχουν τις πληροφορίες για να ανακαλύπτουν, να αποκαλύπτουν και να διορθώνουν τα σφάλματα και μπορούν να τα μειώσουν στο 2%. Ευχαριστώ κύριος Σούλικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ελεγκτικό συνέδριο ακόμη μια φορά βρήκε λάθη τάξεως δισεκατομμυρίων για δέκατο συνεχές έτος Βλέπουμε ότι υπάρχουν λάθη, το διαπιστώνουμε και δεν διορθώνεται τίποτα. Αυτά τα λάθη αφορούν δαπάνες και παραβίαση κανόνων. Παρατηρούμε ότι η πρώτη απέτηση είναι να δαπανηθούν τα χρήματα, δεύτερον να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τρίτον μόνο να δούμε αν έχει νόημα η δαπάνη. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι αυτή η βάση της Ευρώπης να συλλέγουμε χρήματα από τους φορολογούμενους και να τα αναδιανέμουμε. Δεν είναι αυτός ο στόχος της Ευρώπης. Δεν είμαστε Αγιοβασίλειδες. Πρέπει να περικοπούν οι δαπάνες. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι που το κληρονομήσαμε από το παρελθόν, από τον περασμένο αιώνα. Πρέπει να σταματήσει πια. 50 δισεκατομμύρια μας τρώει. Ο κύριος Ζεντεχόφσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, θέλω να σα πω κάτι για την ετησία έκθεση του Ευρωπαϊκού Λευνικού Συνεδρίου. Είναι θλιβερό αυτό το οποίο λέμε εδώ και που προκύπτει σαφώς από την έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από κακή διαχείριση. Ένα σύνδρομο κακή διαχείριση πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και στη νέα θητεία μα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από αυτήν την μάστιγα. Υπάρχει εδώ ένα πολύ βασικό πρόβλημα ότι δηλαδή δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιε είναι οι προτεραιότητέ μα. Όταν λοιπόν γίνεται η δαπάνηση των ευρωπαϊκών πόρων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι πορεία αυτοί δαπανώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κάτι το οποίο προς το παρόν δεν το κάνουμε αρκετά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση το ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτεί ο προϋπολογισμός κατατείνουν να πετύχουν τους στόχους που έχουμε θέσει. Και θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και εσωτερικοί έλεγχοι, θα πρέπει να υπάρχει ακυρεότητα, θα πρέπει να μην υπάρχουν ασυνέπειες. Αυτά είναι τα στοιχεία ε, μιας κακής ε, διαχείρισης. Και τα κρατημέλη επίσης θα πρέπει να δίνουν τα σωστά στοιχεία, άλλοι το κάνουν επίτηδες, άλλοι από ανοργανωσιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν. και τώρα για ένα λεπτό έχει το λόγο κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου για την τόσο πλήρη σας έκθεση. Ας μην ξεχνούμε ότι για άλλη μια φορά το ελεκτικό συνέδριο επισημαίνει τα ίδια και τα ίδια το υψηλό ποσοστό λάθος, το 4,7% το 2013, γιατί είδαμε τι θα γίνει με την ευθύνη όσον αφορά τις δαπάνες των προγραμμάτων αυτό. Είναι κάτι που το έκαναν τα κράτη-μέλη, άρα θα πρέπει εμείς να σκεφτάσουμε εις βάθος γιατί έχουμε τέτοιο ποσοστό λάθος. Να το ψάχνουμε σε βάθος γιατί οι διορθώσεις δεν έχουν αποδώσει όπως θα έπρεπε. Θα πρέπει να εξορθολογήσουμε τους σχετικούς μηχανισμούς, τους μηχανισμούς δαπάνησης, όπως προτείνει το Ελληνικό συνέδριο. Να δούμε επομένως πώς θα πιάσουν τόπο αυτές οι δαπάνες και γιατί θα πρέπει να μην υπάρχει μεταξύ δεσμεύσεων και πληρωμών αυτό το χάσμα. Γιατί οι οφειλές, ε, οι περίμενες οφειλές έχουν επιπτώσεις και για το μέλλον. Οπότε για όλα αυτά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά και εντάχει και θα πρέπει να θεωρήσει ότι αυτά όλα είναι προτεραιότητα υψίστη. Κυρία Σούλη. Α, δεν τη βλέπω, αποσιάζει, οπότε θα πάρει το λόγο μέσα ο κύριος Βάντε Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ε, μικρόφωνο παρακαλώ κύριε Βάντε Δουλεύει, ωραία. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου και την Επίτροπο ε, για τα λεγόμενά τους. Δεν θα σας εκπλήξει ότι θα συμφωνήσω με τον επικριτικό τόνο της κυρίας Γκρέσλε. Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Το ποσοστό των σφαλμάτων πέφτει από 4,8% σε 4,7%. Με κάθε σεβασμό που σας οφείλω, αυτό δεν αρκεί στον Ευρωπαίο πολίτη. Δεν του φτάνει. Ε, δηλαδή δεν πάμε μακριά με αυτό για να το πω λαϊκά. 7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε χάσει. Διαφωνώ σίγουρα με τους συναδέλφους που λένε ότι τα λεφτά πήγαν στη μαφία. Αλλά αυτά τα χρήματα θα πληρώναμε ε, τα, μισά από όσα καθυστερούν για ε, τα, γερμανικά έργα υποδομής. Τι θα κάνετε τα επόμενα χρόνια και ποια διαβήματα προς τα κράτη-μέλη, γιατί αυτά παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι εμείς πιστεύουμε. Και σας ζητώ και πάλι την προσοχή σας, το κάναμε και στις ακροάσεις. Υπάρχουν οι δηλώσεις διαχείρισης των κρατών μελών. Έχουν μεγάλη ευθύνη τα κράτη-μέλη στις δαπάνε και μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύουμε στις Βρυξέλλες. Και τέλος, Πρόεδρε, τι γίνεται με την απλοποίηση και στις αιτήσει και στους λογαριασμούς μπορεί να γίνουν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάμπ. Έχετε μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Χωρί μικρόφωνο κύριος Βαντεκάμπ. Α, από τον κύριο Γκάιερ. Παρακαλώ, 30 δεύτερα. Έχετε μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, αγαπητέ συνάδελφε Βαντεκάμπ, σας ξέρω σοβαρό συνάδελφο εγώ. Γι' αυτό ζήτησα το λόγο, διότι πιστεύω ότι ε, κάνατε ένα λάθος. Είπατε ότι 7 δις χαθήκανε. Να σας διαβάσω τι λέει το ελεκτικό συνέδριο. Το ποσοστό σφάλματος δεν έχει να κάνει με απάτη, με ε, διασπάθηση και Είναι χρήματα που δεν έχουν καταβληθεί. Θα μπορούσα να αποσύρετε αυτό που είπατε ότι έχουν χαθεί 7 δις. 32. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την ερώτηση αυτή. Ε, μπράβο, για να διευκρινίσω αυτά που είπα. Έχει δίκιο, τα 7 δισεκατομμύρια δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά έχουν δοθεί σε λάθος χέρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στο Catch the Eye. Η κυρία Άντερσον πρώτη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ε, ελεγκτές για την δουλειά τους που κανείς δεν την εκτιμάει όπως θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότεροι συνάδελφοι εδώ για τη συζήτηση. Δείχνει η τελευταία του έκθεση πόσο σημασία έχει ο έλεγχος. Να μην ξεχνάμε το βασικό θέμα της απορρόφησης, της χρήσης των πόρων η σωστή απορρόφηση είναι κλειδί. Στην πραγματικότητα γενικά όλα τα χρήματα, πολλά από τα χρήματα που δαπανούμε, βοήθειες για τις πλημμύρες και τα λοιπά, θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί πολύ καλύτερα καθώς και τα ταμεία που στοχεύει συγκεκριμένα η έκθεση. Για να απαντήσω στον συνάδελφο από εκεί πέρα, απέναντι, υπάρχει κατασπατάληση χρήματος αλλά παρακαλώ συνάδελφε τελειώνετε γιατί έληξε ο χρόνος σας. Ο κύριος Μαριάς. Ένα λεπτό επίσης. Η υποκρισία περισσεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ως μέλος της Τρόικας κουνά το δάχτυλο στην Ελλάδα και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και απαιτεί μια βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων με τη δικαιολογία ότι δήθεν είναι ανεπαρκής ενώ η ίδια η επιτροπή δεν μπορεί να βάλει τάξη στα του οίκου της και να ελέγξει τους ίδιους τους υπαλλήλους της για περιπτώσεις ανεπαρκούς δημοσιονομικής διαχείρισης που ρητά αναγράφονται στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώθηκαν αχρεωστήτως, τι θα πείτε κύριοι της Επιτροπής στα εκατομμύρια των ανέργων του Ευρωπαϊκού Νότου για τα σκάνδαλα που περιγράφονται στην έκθεση, για τη διαφθορά στην ανάθεση έργων, για την κατασπατάληση πόρων για την κακοδιοίκηση για το πώς θα πιάσουν τόπο οι δαπάνες δεν είναι λοιπόν δικαιολογημένη και ικανοποιητική η δημοσιονομική διαχείριση εκ μέρους της επιτροπής είχαμε παραβιάσεις κανόνων και πληθώρα σφαλμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σολτές για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και να την καλωσορίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ στο θεσμικό μας όργανο να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Να βλέπουμε αν πιάνουν τόπο με λίγα λόγια είναι γεγονό ότι μπορούν να δαπανούνται καλύτερα, όπω είπε και το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν αμφιβάλλει κανεί γι' αυτό. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και σαφεί στόχου. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό θα πρέπει να μα ενδιαφέρει και εκεί να εστιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επικεντρώσει την προσπάθειά τη. Είναι πολύ περίπλοκοι κανόνε. Δημιουργούν πολλά εμπόδια και δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων αυτών. Υπάρχουν και καλοί κανόνες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έχουν το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο κύριος Έθριτζ, ένα λεπτό. Thank ευχαριστώ. Εγώ εργάζομαι σε Επιτροπή την Περιφερειακή και τώρα έχουμε μελετήσει αυτού του είδους τις ασυνέπειες της ιστορίας και νομίζω ότι δεν πρόκειται για κάτι το δόλιο. Ε, είναι αυθεντικά σφάλματα άρα Σημαντικό να βρούμε μία μέθοδο, ούτως ώστε το σύστημα να μας επιτρέπει μία καλύτερη κατανόηση. Ο κόσμος να μην μπερδεύεται, γιατί τελικά τα περισσότερα λάθη ε, σε αυτό οφείλονται. Πρόκειται για ε, παρανόηση. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται, οπότε θα μπορούσαμε φυσικά να έχουμε παράθυρα μέσω των οποίων έχουμε απάντες και απάντες πολλές εφόσον ε, βρισκόμαστε σε συγκυρία κρίση και όλοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν του λίγου πόρου σωστά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ούτω ώστε τα χρήματα να πιάνουν τόπο και επίση ε, στην διαδικασία δαπάνηση να μην έχουμε σφάλματα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, είπατε επιλέξει ε, ότι η πολίτες περιμένουν από εμά, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επιδείξει ότι ε, δαπανά σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη. Μπορούν να πιστεύουν οι πολίτες τέτοια πράγματα όταν ε, ηγείται της Επιτροπής σας ένας κύριος ονόματι Γιούνκερ, ο οποίος έχει κάνει μυστικές συμφωνίες από ό,τι αποκαλύφθηκε με πολυεθνικές όταν ήταν υπουργό Οικονομικών για να μπορούν να φοροαποφεύγουν όσο θέλουν. Αυτά αφαίρεσε ανίποτα χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς μπορείτε να εμπιστεύεστε ένα τέτοιο άνθρωπο. Οι πολίτες μπορούν να τον εμπιστεύονται. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να παραιτηθεί. Πρόεδρος διακόπτη την ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο έχει τώρα το λόγο. Σε αυτή την ετήσια έκθεση είδαμε τι γίνεται με τις δαπάνες. Το συνεδρίο μας επεσήμανε ότι 2007 με 2013 τι προτεραιότητα δόθηκε στην ε, ε, ποσότητα των εκταμιευμένων και όχι τόσο πολύ στα αποτελέσματα των επιπτώσεων. Πραγματικά έχουμε περίπου ένα μεγάλο ποστό σφάλματος, ε, είπαμε για όλη την περίοδο για 7 δις. Όμως κυρία Γεωργίευα, αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό μου άρεσε ότι δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, να έχουμε ειδικού μηχανισμούς για τις δαπάνες και το ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα. Επίσης θα ήθελα να προσέξουμε το πώς θα περικόψουμε την γραφειοκρατία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτά που λέει το Ευρωπαϊκό Συνέδριο, να είναι πιο ρεαλιστική όσον αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, όπως κάθε Χριστούγεννα, κάθε χρόνο έρχεται ο Άγιος Βασίλης, το ελεκτικό συνέδριο. Τι ε, ωραίο υλικό μας δίνουν και ευχαριστούμε. Αλλά δεν είναι συνταρακτικά αυτά. Εδώ και πέντε χρόνια τα ίδια ακούω. Τις προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που ε, συστηματικά αγνοούνται. Κάνετε και καλές προτάσεις για την πρακτική ε, εφαρμογή και την πρακτική χρησιμότητα. Δεν θα πρέπει να γελιόμαστε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πραγματικοί στόχοι δεν είναι προτεραιότητα όμως, ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, με άσχετα. Πού είναι ε, τα θέματα, η προστασία του περιβάλλοντος λέει προστασία των ζώων και κάτι τέτοια. Η Ένωση μου θυμίζει ένα πολύ βαρύ δεξαμενόπλιο γεμάτο πετρέλαιο που πάει ε, προς ολοταχώς και άμα του συμβεί κάτι δεν μπορεί να στρίψει. Ε, και έχει και ένα καπετάνιο που δεν θέλει καν να αλλάξει ρότα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γεωργίευα, παρακαλώ, έχει το λόγο. Thank you, madam. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να αρχίσω με ευχαριστίες για τις παρατηρήσεις. Τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα. Πάρα πολύ ευχαριστώ και όλοι εκείνοι οι οποίοι είπαν ότι επιθυμούν να έχουμε καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση προς χάρη των Ευρωπαίων Έχω να σας αναφέρω τρία τινά. Πρώτα πρώτα, τι ακριβώ σημαίνει ποσοστό σφάλματος. Το εξή. Λάθη, σφάλματα. Ορισμένα από λάθος διαχείριση των πόρων, αλλού έχει γίνει λάθος στην εγγραφή των ε, κονδυλίων και ένα 0,2% ένα μικρό ποσοστό είναι χρήματα τα οποία υπεξερέθηκαν. 0,2% είναι 0,2% είναι κάτι. Είναι πολύ. Όμως δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε τα ασφάλματα τα οποία πραγματικά είναι υλικά, υλικού πρακτικού χαρακτήρα με την κακοδιαχείριση ή με την απάτη. Θα πρέπει η διάκριση να είναι σαφής. Θα πρέπει να περιχαρακώσουμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το επιλύσουμε. Δεύτερον, τι κάνουμε για το πρόβλημα αυτό. Για τα περισσότερα σφάλματα που είναι αυτό που λέει η λέξη σφάλματα με τα κράτη-μέλη ακάματα προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε στελέχη που ασχολούνται με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Και διαπιστώνουμε ότι αξίζει της προσοχής μας αυτή η προσπάθεια. Γιατί Εάν έχουμε κάποιους οι οποίοι αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν τις διατάξεις, τότε συρρυκνώνεται το ποσοστό σφάλματος και έχουμε πολλές ενδείξεις ότι τέτοια προγράμματα κατάρτισης οδηγούν σε μείωση του ποσοστού σφάλματος και όταν δεν κάνουμε αυτό, αντιθέτως, ε, εκτινάσεται στα ύψη αυτό το ποσοστό σφάλματος. Άρα αν έχουμε στη νέα περίοδο προγραμματισμού κάποιο είδους ε, κίνητρα, δηλαδή 6% των χρημάτων αποτελούν αποθεματικό ούτω υπήν με το οποίο να μπορέσουμε να αμύψουμε τις καλές επιδόσεις, να έχουμε και αντικίνητρα, να έχουμε δηλαδή κάποιο είδου κόψιμο των πόρων εκεί που θα υπάρχει κακική διαχείριση των κοινωνικών πόρων. Οπότε κάνουμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα και να πλουστεύσουμε τις διατάξεις και τους κανόνες. Έχουμε τώρα διατάξεις σχετικές με την επιλεξιμότητα, θέλουμε να γίνει εναρμόνιση για πολλούς τομείς, όμως θέλω να σας πω κάτι. Χθες Μίλησαμε για δαπάνε με του ανθρώπους στην Επιτροπή για να δούμε τι γίνεται, πώ μπορούμε το θέμα αυτό να το προωθήσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω τα είπε το Ελληνικό Συνέδριο. Το τρίτο που θέλω να σα πω είναι Παίρνουμε στα σοβαρά την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Η απάντηση είναι καταφατική. Τι μα είπε το Ελληνικό Συνέδριο, έκανε στην ε, ε, έκθεση ειδική έκθεση 19 του 2013, ότι θα πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη οι συστάσεις και ότι έγινε μια αναθεώρηση αυτών των παλαιότερων συστάσεων και θεώρησε ότι βελτιώθηκε η διαχείριση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη αυτές τι συστάσει. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να πάρουν πάρα πολύ σοβαρά και ιδίως όσον αφορά την στροφή που θα πρέπει να κάνουμε, όσον αφορά ε, την αυστηρή συμμόρφωση ε, προς το πώς θα έχουμε μία, πώς θα δώσουμε την έμφαση, πώς θα προσέξουμε περισσότερο το αποτέλεσμα της τελικές επιδόσεις. Ελπίζω ότι του χρόνου θα έχουμε κάποια αποτελέσματα καλύτερα να τα συζητήσουμε. Και εγώ σας ε, υπόσχομαι ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα προς το καλύτερο να συζητήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ο κύριος Σίλβα Καλντέρα για να ολοκληρώσει συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα καλά τους λόγια προς το ελεκτικό συνέδριο και σας ευγνωμονούν όλοι όσοι συμμετείχαν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Τα αγγλικά τώρα θα ήθελα να απαντήσω σε πολλά από τα σημεία που ανέκυψαν στη συζήτηση. Όχι επειδή απευθύνεστε σε εμά προς απάντηση, αλλά γιατί πρέπει να έχουμε σαφή ιδέα για το τι ε, δέον γενέστε. Στην έκθεσή μας εμείς ρητά αναφέρουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, αυτή η κουλτούρα, ότι χρησιμοποιούμε τα λεφτά γιατί υπάρχουν. Αλλιώς θα τα χάσουμε. Ε, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα δαπανίσουμε. Θα πρέπει τα συστήματα να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Είδαμε και δείξαμε στην έκθεσή μας ότι τα κράτη-μέλη έχουν την πληροφόρηση για να ε, ε, τα ζητήσουν και να ε, μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Θέλουμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν ακριβώς τη δουλειά τους για να αυξηθεί αυτή η προληπτική δράση. Βεβαίω, σφάλματα γίνονται, άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Αλλά ε, αυτά θα πρέπει να διορθώνονται και να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος της διορθωτικής δράσης και της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Τελικά, σε κάποιους τομείς, ακόμα και έτσι, και σε κάποιες ε, περιπτώσεις που ελέγξαμε, καταφέραμε να μειώσουμε ε, το σφάλμα ε, πολύ κοντά ε, στο αποδεκτό. Λοιπόν, οι κανόνες είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται να αλλάξουν και πάλι για τη νέα προγραμματική περίοδο. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα τελικά είναι η εφαρμογή. Ζητήσαμε να αλλάξουμε τους κανόνες, τους αλλάξαμε. Τώρα έχει έρθει η ώρα της δράσης. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβουν τώρα τη δράση. Με την απλούστευση, την απλοποίηση των κανόνων και με την σωστή στόχοθεσία με τα σωστά προγράμματα που είναι σχεδιασμένα ε, και στραμμένα στα αποτελέσματα για να έχει αυτό πραγματικό αντίκτυπο στις ζωές των ε, Ευρωπαίων πολιτών αλλά με τα σωστά κίνητα. Και εκείνα με τις καλύτερες επιδόσεις θα πρέπει να πρημοδοτούνται. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κλείνοντας να επαναλάβω ότι αυτή, αυτή η νέα εστίαση ε, που πλέον στοχεύει σε ορατά αποτελέσματα για τους πολίτες θα πρέπει να είναι ο ακρογωνίος για το μέλλον. και έτσι θα έχουμε ευημερία, απασχόληση στην Ευρώπη και θα έχουμε και τελικά και προστασία του περιβάλλοντος. Ε, όλοι προς αυτή την κατεύθυνση κοιτάμε. Ε, και απευθύνομαι και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί σε εκείνη αναπόκειται και στα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν σε αυτά τα θέματα. Και σε αυτή την κουλτούρα και την οτροπία. Όταν έχουν χρήματα της Ένωσης να δαπανίσουν να κοιτούν για ποιο αποτέλεσμα και όχι απλώς να τα απορροφήσουν. Ευχαριστούμε κύριε μου. Λίγη αυτή η συζήτηση και τώρα προβλέπεται η δήλωση της Επιτροπής για την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Χαίρετε κυρία Γεωργίευα. Ναι.